την έγκριση των πρακτικών οι αλλαγές αυτές θα θεωρηθούν εγκριθήσεις. Η δεύτερη ανακοίνωση είναι η εξής. Σύμφωνα με το κανόνα 152 εδάφιο 2 και σύμφωνα με και σε συμφωνία με τις πολιτικές ομάδες σας προτείνω την εξή αλλαγή στην ημερήσια διάταξη τη Τετάρτη. Η συζήτηση για το προφορικό ερώτημα προ το Συμβούλιο και την Επιτροπή για την παρακολούθηση τη συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου τη 11 11 Φεβρουαρίου του 2015 για την έκθεση της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών για την χρήση των βασανιστήριων από τη CIA πρόταση είναι να αναβληθεί για να εκπροσωπηθεί αρμοδίως στο Συμβούλιο γιατί πρέπει το Συμβούλιο να αποχωρήσει απόψε το βράδυ. Ε, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, τροποποιείται η μερίσια διάταξή μα αναλόγω. Ευχαριστώ. Ερχόμαστε τώρα στι ψηφοφορίε. Πρώτη έκθεση είναι η έκθεση Χαουτάλα προστασία έναντι των επιδοτούμενων εισαγωγών από χώρες.